Ε, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επαναλαμβάνω, λάβατε θέσεις. I would like to continue. Θα συνεχίσουμε με βάση αυτά που είπε ο Αντιπρόεδρος Μαρτίνες πριν από λίγες ώρες. στην Ισπανική επαρχία της Μούρθια έγινε σεισμός. Σκοτώθηκαν τουλάχιστον 8 άνθρωποι, υπάρχουν πολλοί τραυματισμένοι και ανακοινώθηκε πριν από τρεις ώρες από τον Αντιπρόεδρο Μαρτίνες το νέο. Θα ήθελα εξ ονόματος του Κοινοβουλίου να εκφράσω τα συλληπιτήρια για τα θύματα και τις ευχές μας για σύντομη θεραπεία και ίαση των τραυματιών. Θα στείλουμε συλληπιτήριο τηλεγράφημα στην Ισπανική κυβέρνηση. Η Χριστίνα Γκουτιέρες ή ο κύριος Μαρτίνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα καλά σας λόγια ένδειξη Τσιμπονιές και αλληλεγγύης. Η τραγωδία της ε, Λόρκα αναπτύσσεται. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή 8 θανάτους, μεταξύ των οποίων 3 έγκυες γυναίκες και ένα παιδάκι 8 ετών. 80% των ε, κατοικιών έχουν ε, πληχθεί. Από εδώ και πέρα λοιπόν νέα τους κατοικία θα είναι ο ουρανός υπάρχουν και άνθρωποι που έχασαν το χώρο εργασία τους, ε, ε, έχασαν τις ελπίδες τους, ε, τις προσδοκίες τους και τις ευκαιρίες τους. Η Λόρκα είναι μια πόλη 70.000 κατοίκων με πάρα πολλούς μετανάστες, τους οποίους δέχτηκε, υποδέχτηκε και τους έδωσε μια νέα ζωή και νέο νόημα. Μαζί, λοιπόν, παλιοί κάτοικοι και νέοι κάτοικοι με τη βοήθεια όλων των θεσμικών οργάνων θα μπορέσουν ίσως να ξαναξεκινήσουν τη ζωή τους. Αλλά Πρέπει να πω ότι η Ευρώπη δεν θα πρέπει να αφήσει κανέναν πίσω και ξέρει να γνωρίζει αυτούς που πάσχουν. Να, να γνωρίσει που υπάρχει ο πόνος και να τους ε, υποδεχθεί με ανοιχτές αγκάλες. Ευχαριστώ σε όλους και θα ήθελα να ζητήσω ένα λεπτό ε, Ευχαριστώ. Θα τηρήσουμε τώρα ενός λεπτού σιγής.